Uh, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα Σας παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις σας επειδή με ιδιαίτερη χαρά έχουμε υποδεχθεί τον Κάρελ Ντεγκούχτ ο οποίος έχει έρθει για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό θα ήθελα να αρχίσουμε αν δεν έχετε αντίρρηση και βεβαίως τα επόμενα λεπτά θα έρθουν και άλλα μέλη. Θα ήθελα να εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη, εάν συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του Προέδρου. Υπάρχουν τα πρακτικά της 26 Οκτωβρίου που μπορούμε να τα εγκρίνουμε εκτός αν υπάρχουν παρατηρήσεις με, τη συνήθεια διαδικασία. Ο κύριος Ντεγκούχτη είναι εδώ για να απαντήσει σε ερωτήσεις μας. Τον υποδεχόμαστε με χαρά στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς διότι παρόλο που δεν έχουμε νομοθετικό έργο με εσάς, σε συνεργασία με εσάς, η Επιτροπή μας ε, ε, παρακολουθεί τις επιπτώσεις τις ευρύτερες επιπτώσεις στην ε, εσωτερική, για την εσωτερική αγορά για τα θέματα της τυποποίησης κλπ. Οπότε υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνουν οι υπηρεσίες σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε την πρόσκληση να έρθετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες για όλα αυτά τα θέματα. Επειδή πρόσφατα επιστρέψαμε από μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή στην Ινδία, πριν από δύο χρόνια είχαμε πάει στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε επίσης και όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε αναλάβει με πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ ευτυχείς που είστε εδώ. Με τα χαρά θα σας δώσω το λόγο και μετά θα δεχθείτε ερωτήσεις από τα μέλη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου ενέκρινε την, ανακοίνωσή ε, ε, της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της εμπορικής πολιτικής, εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις. Έδωσα στην Επιτροπή μια σύντομη ε, επισκόπηση των κύριων σημείων της ανακοίνωσης σήμερα και χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να κάνω το ίδιο με τη δική σας Επιτροπή λόγω της σημασίας που έχουν οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές μας, οι οποίες είναι αλληλένδετες. Θα μιλήσω για την τυποποίηση σε λίγο και το ρόλο της ε, αρχίζοντας με την ανακοίνωση, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί ε, και να ανταποκριθούμε σε αυτά που έχουμε ήδη υποσχεθεί, δηλαδή να ολοκληρώσουμε τα επόμενα χρόνια μια σειρά από φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες σε πολυμερές επίπεδο και σε διμερές επίπεδο με αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες σε κάθε γωνιά της γης. Δεύτερον, πρέπει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας, τις εμπορικές μας σχέσεις με άλλους μεγάλους εταίρους, την Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ιαπωνία και να προωθήσουμε συζητήσεις για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και συμπράξεις προωθώντας ε, τις επενδύσεις και την κατάργηση των ε, εμποδίων στο εμπόριο. Και ε, σε αυτό το τομέα προσβλέπουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή σας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ορισμένα φόρουμ όπως το οι με τις Ηνωμένες, το, Συμβούλιο με τις Ηνωμένε Πολιτείες θα ορίσουν, ορίσουν τις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες και θα επιλύσουν προβλέποντάς, τις, προβλέποντάς τα ε, ρυθμιστικά προβλήματα με νομοθεσία για διάφορους τομείς. Και ε, η Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή ΙΜΚΟ θα θεσπίσουμε ορισμένους κανόνες. Τρίτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν όλοι για να προωθήσουμε την απασχόληση για την προώθηση εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί πρέπει να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Τέταρτον, οι ξένες επενδύσεις είναι μια κινητήρια δύναμη για επενδύσεις και ανάπτυξη. Πάρα ε, πολλά εκατομμύρια εργάζονται και μόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κινέζικες και άλλες ξένες εταιρείες. Προτείνουμε λοιπόν μια πιο επιθετική προσέγγιση στην ε, ε, εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών προστατεύοντας τα δικαίωματά μας και εξασφαλίζοντας ότι ισχύουν για όλους οι ίδιοι κανόνες. Θέλουμε η εμπορική πολιτική μας να προσφέρει ωφέλη μακροχρόνιας ανάπτυξης και μεγαλύτερης ευημερίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρώπη απορρίπτει τον προστατευτισμό και πρέπει να ενεργούμε κατά των προστατευτικών μέτρων που λαμβάνουν οποιασδήποτε χώρε. Από την άποψη αυτή, οι δεσμεύσει που ανέλαβε το G20 στη Σεούλ θα δώσουν νέα όθηση σε αυτές τις προσπάθειες. Τέλος, το εμπόριο πρέπει να είναι συμμετοχικό ώστε όλοι να απολαμβάνουν τα ωφέλη της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό ισχύει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμα περισσότερο ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου το εμπόριο να χρησιμοποιηθεί σαν ε, στήριγμα για ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην παγκόσμια αγορά. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για την τυποποίηση. Χαιρετίζω τις, τις εκθέσεις σας για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης με πρωτοβουλία του Έντβαρ Κρατζίτσκι που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διαδικασία της τυποποίησης είναι ευθύνη του Αντώνιου Ταγιάννη, του συναδέλφου με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε σε όλα τα επίπεδα. Στις αρχές του 20ου ε, αιώνα, τα του 21ου αιώνα, δημιουργούνται νέα πρότυπα διότι υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί η διασύνδεση ανάμεσα στις τεχνολογίες μειώθηκαν, μειώθηκε η χρήση εταιρικών και εθνικών προτύπων που αντικαταστάθηκαν από διεθνή πρότυπα. Ένας από τους λόγους για την εξέλιξη αυτή είναι η συνεχιζόμενη, το, συνεχιζό, το αυξανόμενο διαρκώς διεθνές εμπόριο. Η τυποποίηση παίζει σημαντικό ρόλο διότι αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και είναι σημαντικό μέσο για την κατάρτιση των εμπορικών εμποδίων και την προώθηση των εμπορικών ρευμάτων. Τα μη δεσμολογικά εμπόδια και η προώθηση των προτύπων έχουν μεγάλη σημασία για τις σχέσεις μας με άλλους εταίρους και έχουν θεωρηθεί ως οι βασικότερε προκλήσεις στην ανακοίνωση για το μέλλον της εμπορική πολιτικής. Ρυθμιστικά εμπόδια στο εμπόριο και στις υπηρεσίες και τι επενδύσει έχουν ζημιογόνε επιπτώσεις στις σχέσεις με τους κυρίους εμπορικούς εταίρους μας λόγω των σχέσεων που διατηρούμε με αυτούς συνεργασία στον τομέα των ρυθμίσεων είναι αναγκαία για να προωθηθεί η σύγκληση, η, ισο... Ε, η αντιστοιχία των κανόνων και των πρακτικών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε ε, δυνητικά εμπόδια προτού ευδρεωθούν ορισμένες ρυθμιστικές διατάξεις έχουμε ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Κίνα, προωθώντας την καθιέρωση διεθνών προτύπων. Η διεθνής τυποποίηση είναι ένα σημαντικό θέμα που συζητείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνής τυποποίηση είναι ένας τρόπος να ξεπεραστούν τα εμπόδια σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η έκδοση η εξασφάλιση ε, πιστοποιητικών που χορηγούνται από το Διεθνό Οργανισμό Τυποποίηση, την Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή, την Ένωση Τηλεπικοινωνιών και την ε, Επιτροπή του ΟΗΕ για τα οχήματα έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμα το Ιδιατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο που είναι η κυρίως πλατφόρμα για την οικονομική ρυθμιστική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό σε ορισμένου τομεί όπω είναι η βιοτεχνολογία ή οι υπηρεσίε online. Πρέπει να προωθήσουμε τι ε, προσπάθειές μας σε άλλους τομείς όπως τα χημικά προϊόντα θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστές. Ανταγωνιστικοί πρέπει με ρεαλισμό να αντιληφθούμε ότι η προσέγγιση μας για τα πρότυπα και η ευρύτερη προσέγγιση μας στις ρυθμίσεις θα παραμείνουν διαφορετικές αλλά πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να προσπαθούμε να, κάνουμε, να πετύχουμε κάτι το καλύτερο αποφεύγοντας ε, τριβές και προβλήματα. Γι' αυτό εστιαζόμαστε σε συνεργασία μεταξύ, Ευρωπαϊκής, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ και μεταξύ νομοθετών. Χρειάζεται η αντίστοιχη προσέγγιση για την Ιαπωνία, με την οποία έχουμε εντείνει το διάλογο για τα τεχνικά εμπόδια που παρεμποδίζουν τις διμερείς εμπορικές μας σχέσεις. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της ομάδας υψηλού επίπεδου η οποία έχει αναλάβει το έργο να, να... Ε, ε, να δείξει με ποιους τρόπους θα βελτιώσουμε τις, εμπορικές, τις διμερείς μας σχέσεις. Στα... Ε, Στι εμπορικέ συμφωνίε που έχουμε ήδη υπογράψει, έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στη χρήση των διεθνών προτύπων, ενισχύοντα την εργασία σε αυτό το τομέα. Επιπρόσθετα, τις συμφωνίες για τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις από, μετά από την ανακοίνωση του 2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διευρύνει το, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σε, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τις ρυθμίσεις στην ε, πρόσφατη συμφωνία με την Κορέα εξασφαλίσαμε από την Κορέα τη δέσμευση ότι θα εφαρμόζει ορισμένα διεθνή πρότυπα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα δέχεται για ηλεκτρονικά προϊόντα ε, πρότυπα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόοδο της ευρωπαϊκής τυποποίησης και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό τον τομέα. Επειδή η σύμπραξη με τους νομοθέτες θα είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη μας για ερωτήσεις. Είμαστε πολύ ευτυχής που η εργασία που κάναμε έχει εκτιμηθεί από τον Επίτροπο. Ξέρω ότι τα, τα περισσότερα μέλη μας θα ήθελαν να θέσουν ερωτήσεις. Η κυρία, ο κύριος Σβάμπ, ε, η κυρία Βάιλερ, η κυρία Κόζουτσνικ. Δίνω λοιπόν καταρχάς ε, το λόγο για τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Θέλετε να απαντήσετε ομαδικά σε μερικές ερωτήσεις μαζεμένες ή... Ωραία, ειδικά για το θέμα της τυποποίησης. Ο κύριος Σβάμπ, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε στην Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς και νομίζω ότι ήταν λίγαν κατάλληλη εποχή που σας κάλεσε η Επιτροπή μας βάσει όλων όσων διαβάσαμε στο, στην έκθεση του Επιτρόπου Μόντι. Η εσωτερική αγορά και η προστασία των καταναλωτών θα γίνει ένα θέμα όλο και μεγαλύτερης σημασίας. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι οι κανόνες του εμπορίου πρέπει να ισχύουν για όλους. Σε αυτό συμφωνούμε και όλοι πρέπει να σας υποστηρίξουμε στην ε, ε, εφαρμογή αυτής της αρχής. Αλλά δυστυχώς δεν ισχύει αυτό στην πραγματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται στην κατασκευή των, πολωνικών αυτοκινήτων δρόμων. Και είδαμε ήταν ένα κακό παράδειγμα διότι δεν υπήρχε μία ισότιμη διαδικασία μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού και έτσι δεν μπόρεσαν πολλά από τις, πολλές από τις εταιρείες μας να λάβουν μέρος στην ανάθεση. Όταν κοιτάξουμε την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της εσωτερικής αυτής αγοράς στους πολίτες μας, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όταν, παραδείγματος χάρη, <clears throat> ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όχι του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στους δημόσιους διαγωνισμούς τρίτων χωρών και έτσι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων εταιριών που χαίρουν κρατικές επιδοτήσεις. Το έχω συζητήσει αυτό με τον Ντάνιελ Κασπάρη στο παρελθόν από, στην Επιτροπή Εμπορίου και θα συζητήσαμε κατά πόσον οι κανόνες του GPA θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλλον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει μια πιο ισότιμη, όπως θέλετε και εσείς, ίση μεταχείριση. Μια θεμελιώδης αρχή, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει. Η κυρία Γκέπαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις Δύο σημεία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Το πρώτο σημείο το ανέφερε ήδη ο κύριος Σφάμπ και είναι η ισότιμη μεταχείριση στην παγκοσμιοποιημένη αγορά στην, ε, στον τομέα του εμπορίου, των εμπορικών συναλλαγών. Έχω όμως και μία ακόμα ερώτηση. Ωραία είναι να λέμε ότι όλοι θέλουμε ισότιμη μεταχείριση, ισότιμους κανόνες, έτσι ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά. Αλλά σε ποιο επίπεδο, για ποιο επίπεδο μιλάμε, δηλαδή σε ποιο επίπεδο θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή την ισότητα, την ισονομία. Εμένα με ενδιαφέρει το θέμα από κοινωνικής απόψεως. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω όταν υπογράφει συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή πώς λαμβάνεται υπόψη αυτό το θέμα το, της κοινωνικής διάστασης και σε ποιο επίπεδο θέλετε να εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις. Δεύτερον, όταν κλείνονται εμπορικές συμφωνίες κατά πόσον είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, την υλοποίηση ε, έχω ακούσει τελευταίως ότι αυτή την εποχή υπάρχουν τεράστιες ε, δυσκολίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας από την άλλη πλευρά όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα στην υλοποίηση δεσμεύσεων οι οποίες έχουν συνυπογραφεί από τους εταίρους αλλά δεν εφαρμόζονται. Πώς μπορείτε λοιπόν να διασφαλίσετε μια ακριβή εποπτεία των συμφωνιών και εφαρμογή τους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα να απαντήσει ο Επίτροπος σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Όχι, πιστεύω ότι... The uh, Πιστεύω ότι στην, στο ανακοινωθέν στην ανακοίνωση του εμπορίου που έγινε, για, για το, τις εμπορικές συναλλαγές, για το τομέα του εμπορίου που έγινε, έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε όλα αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι τώρα ε, έχουμε ως στόχο οι νομοθετικές μας ρυθμίσεις να έχουν και διεθνείς επιπτώσεις. Δηλαδή να υπάρχει μια διεθνής πτυχή στην νομοθεσία που διέπει το εμπόριο ε, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια αμοιβαιότητα. Θα σας ε, δώσω ένα παράδειγμα όπως και η κυρία Γκέπαρτ ανέφερε συγκεκριμένο παράδειγμα όσον αφορά την αμοιβαιότητα. μια κινέζικη εταιρεία η οποία κατασκευάζει αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρομικά δίκτυα στην Πολωνία και λέγεται, αν και δεν είναι απόλυτα σαφές, ότι δόθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για αυτά τα έργα. Έτσι φημολογείται, το οποίο είναι, ε, ε, είναι προσβλητικό θα έλεγα. παρόλο που μπορεί να μην έχει μεγάλη οικονομική επίπτωση, ε, εάν πράγματι συνέβη, είναι αθέμητος ανταγωνισμός και ε, είναι μια κατάχρηση της ε, ίσης μεταχείρισης. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους παρέμβασης για να μην επαναληφθούν αυτά τα γεγονότα, αυτά τα κακά παραδείγματα. Ε, μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα ή να κλείσουμε τις αγορές, δηλαδή προστατευτικά βεβαίως, με προστατευτικά μέτρα ή να ενισχύσουμε τη θέση μας σε διεθνή ε, στις διεθνείς διαβουλεύσεις, ε, στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, το οποίο βεβαίως εγώ υποστηρίζω Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση που αναφέρατε για τις βόρειες χώρες της Ένωσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις με τη Ρωσία δεν νομίζω ότι έχει απόλυτη σχέση με την εφαρμογή, την υλοποίηση των συμφωνιών. Διότι, όπως ξέρετε, η Ρωσία δεν είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που σημαίνει ότι είναι σε θέση να αυξήσουν τους δασμούς και να επιβάλλουν εξαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα και γι' αυτό είναι προφανές ότι έχουν ακουστεί πολλά αρνητικά σχόλια όμως το πρόβλημα δεν λύνεται με εφαρμοστικά μέτρα. Επειδή δεν είναι μέλη του ΠΟΕ, μπόρεσαν να ε, κάνουν αυτά τα, αυτές τις ενέργειες και γι' αυτό είναι σημαντικό η Ρωσία να γίνει μέλος του ΠΟΕ. Την περασμένη εβδομάδα συνήψαμε μια διμερή συμφωνία με τη Ρωσία για τις προϋποθέσεις ένταξής του στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και χρειαζόμαστε ακόμα να συμπληρωθεί και συμφωνηθεί το πολυμερές κεφάλαιο το οποίο θα ολοκληρώσουμε στη Γενέβη. Εκεί θα γίνουν διαπραγματεύσεις και έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα όπως και τους εξαγωγικούς δασμούς επί της ξυλίας οι οποίοι θα μειωθούν κατά τα 2 τρίτα και μόνο το 1 τρίτον του ύψου των δασμών θα παραμείνει και νομίζω ότι οι βόρειες χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι λίγαν ικανοποιημένες αν επιτευχθεί αυτή η πρόοδος. Ε, στην ανακοίνωση που είπαμε τονίζουμε ότι θα, θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στην υλοποίηση ακριβώς επειδή υπάρχει συμφωνία. Όταν υπάρχει μία συμφωνία δικαιούσε να ζητήσεις και τον σεβασμό των συμφωνημένων ε, διατάξεων της συμφωνίας, ε, του περιεχομένου της συμφωνίας. Η Ρωσία πρέπει να πειθαρχήσει, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν γίνει μέλος του ΠΟΕ και οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε το ταχύτερο να γίνει μέλος για να πειθαρχήσει. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις ε, απαντήσεις σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το, τώρα τον κύριο Σάλντομος και την κυρία Βάιλερ. ο κύριος Λούκεγκαρτ και ο κύριος Έγκστρομ επίσης, αν θέλουν η κυρία Σάλντομαλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και ευχαριστώ και για την παρουσίαση αυτή. Εγώ συμμερίζομαι απόλυτα μαζί σας την άποψη αυτή για τα προβλήματα που μπορούν να τεθούν σε επίπεδο εμπορίου και ως προς τις ενδοκινοτικές και εξοκινοτικές σχέσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την συνοχή. Δηλαδή, πώς συμβαδίζει η δική μας εσωτερική εμπορική πολιτική με την εμπορική ε, πολιτική που έχουμε προς τρίτες χώρες. Εγώ ε, είχα μεταβεί στην Ιαπωνία μέσα στα πλαίσια των διμερών και πολυμερών σχέσεων με την Ιαπωνία και έγινε λόγος για σύναψη εμπορική συμφωνίας με αυτή τη χώρα, αλλά μιλήσαμε και για πιο άμεσες σχέσεις και με τους βουλευτές έφνης από την Ιαπωνία. Δηλαδή να υπάρχει ένας ε, διακοινωτικός διάλογος και από ό,τι είδα δεν υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον από πλευράς ε, Ιαπωνίας. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας από τους Ιάπωνες. Θα πρέπει όμως να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συντονιστούμε και να μην ανταγωνιζόμαστε οι μεν τους δε. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωβουλευτές για να υποστηρίξουμε αυτή την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε στην ΙΜΚΟ για να προωθήσουμε αυτή την εργασία έτσι ώστε να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και όχι αθέμητος μέσα στο πλαίσια του νομοθετικού διαλόγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν, ε, δεν συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη σας απάντηση, κύριε Επίτροπε, διότι όταν απαντήσατε ε, για στο θέμα της ε, Πολωνίας ε, και τους εργαζόμενους από την Κίνα ή την Ουκρανία κλπ. Θέλω να επανέλθω σε αυτό, διότι έχω παρόμοια προβλήματα με τον κατασκευαστικό τομέα στο κρατήδιο της ΕΣΥΣ όπως και οι συνάδελφοί μου. Δεν με ικανοποιεί απόλυτα η απάντηση, διότι πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσουμε. Όταν πρόκειται για επιδοτήσεις πρέπει να ενεργήσουμε. Πρέπει να δράσουμε. Όταν δεν πρόκειται για επιδοτήσεις το θέμα είναι πολύ δύσκολο διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητες ούτε νομοθετικές ούτε οικονομικές μέσω συμφωνιών. Όταν όμως πρόκειται για επιδοτήσεις τις οποίες η Πολωνία λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον στο παρελθόν όταν μαθαίναμε ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί τότε σε κάθε φορά αυτό κόπηκε. Σταμάτησε. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι ένα, μικρό, ένα παράδειγμα ε, με μικρές επιπτώσεις, με περισμένες επιπτώσεις. Αλλά μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Ε, ξέρω ότι πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν παραδείγματος χάρη στην Πολωνία, μετά πάνε στην Ουκρανία και δημιουργούνται παρόμοια προβλήματα από ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν σε ένα τρίτο κράτος και δουλεύουν μια χαρά. Θέλω λοιπόν να ξέρω εάν έχουν δοθεί κονδύλια και η πολωνική κυβέρνηση πρέπει να μας ε, δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες όπως έγινε και στο παρελθόν όταν υπήρχαν παρόμοιες περιπτώσεις. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σήξω είναι η Ινδία και η συμφωνία FTA με την Κορέα και τη Σιγκαπούρη. Είναι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και για μας αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική διότι στην Ινδία μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μας τους ευρωβουλευτές. Δηλαδή δεν θα υπάρξει έλεγχος εάν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε θέσει θα εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την παιδική εργασία στον τομέα της κατασκευής των χαλιών όπου μικρά παιδιά χρησιμοποιούνται επειδή έχουν επιδέξια χέρια Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση και να μην χαθεί η εποπτεία και ο έλεγχος με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα με αυτές τις περιπτώσεις και με τις άλλες χώρες με τις οποίες εσείς προβλέπετε να συνάψετε συμφωνίες. Θα εξετάσετε την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, αυτών των προϋποθέσεων που τέθηκαν, διότι έχει μεγάλη σημασία και τα οικονομικά και τα κοινωνικά κριτήρια να γίνουν σεβαστά και θα ήθελα να ξέρω ε, αν παρακολουθείτε την εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε και πάλι θέση γιατί το μικρόφωνο σας νομίζω δεν λειτουργεί. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Um, Πρώτα, σχετικά με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία μας ζητά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών είχαμε συναντήσει τον περασμένο Μάιο νομίζω με την Ιαπωνία όπου καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε πρώτα να καταργήσουν τα, τα μη εμπορικά εμπόδια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε με την Ιαπωνία. Πολύ περισσότερο από τους δεσμούς είναι το πρόβλημα των μη εμπορικών εμποδίων και έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα εξετάσει όλα τα εμπόδια που υπάρχουν για το εμπόριο και η έκθεσή της θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής με την Ιαπωνία που πρόκειται να λάβει χώρα γύρω στον Απρίλιο του 2011 στις Βρυξέλλες. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Με ρωτήσατε και για τον ανταγωνισμό. Μάλλον αφορούσε ειδικά την Ιαπωνία, ήταν γενικότερη, ε, ευρύτερη ερώτησή σας. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας παραλληλισμός ανάμεσα σε αυτά που κάνουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το υποβάλλετε στον Ιωακή Αλμούνια, διότι ο Επίτροπος Αλμούνια έχει αρμοδιότητα την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης όταν υπάρχει μια σχέση η οποία μας δίνει η οποία μπορεί να εφαρμόζεται και εκτός της επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Κίνα υπάρχουν πολλά προβλήματα διότι στη χώρα αυτή υπάρχουν ε, υπηρεσίες, ε, οργανισμοί που έχουν ορισμένες αρμοδιότητες. Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είναι η κατάσταση με την Ιαπωνία, αλλά νομίζω ότι κάθε χώρα ε, εξειδικεύεται σε μέσα και εργαλεία που θα προστατεύσουν την αγορά της και η Ιαπωνία το κάνει αυτό με μη δασμολογικά εμπόδια. Για την Πολωνία. Δεν ξέρω γιατί δεν σας ικανοποίησε η απάντησή μου. Από τις ερω... Ίσως δεν ήταν ε, απόλυτα σαφής η ερωτήση σας. Αυτό που έλεγα ήταν ότι θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε και να κλείσουμε ορισμένους τομείς ε, σε ό,τι αφορά τις κρατικές προμήθειες και την αγορά των κρατικών προμηθειών. Αυτό πιστεύω που εννοούσατε ήταν ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς, δηλαδή μέσα αμυντικά όπως το αντι και τα εχέγγυα και οι εγγύησει. Αυτό είναι κάτι που πράγματι θα μπορούσε να γίνει, αλλά είναι και θέμα, επίσης θέμα χρονικής συγκυρίας, timing. Προτού ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, πρέπει να ε, υπογραφεί μια σύμβαση. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Για να παρέμβουμε στον τομέα των κρατικών προμηθειών χρειαζόμαστε ένα νέο εργαλείο και θα υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μας εξασφαλίσει αυτό το νέο μέσο, αυτό το νέο εργαλείο που θα ενταχθεί στα διάφορα μέσα προστασίας του εμπορίου που διαθέτουμε. Για την Ινδία τώρα. We are making serious progress. Έχουμε πραγματικά σημειώσει μεγάλες προόδους στις διαπραγματεύσεις μας με την Ινδία. Θα γίνει μια σύνοδος κορυφή με την Ινδία στις 10 Δεκεμβρίου, σε 15 μέρες δηλαδή περίπου. Και αναμένουμε Πρέπει βεβαίως να είμαστε προσεκτικοί, αλλά αναμένουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ιδία μέχρι την επόμενη άνοιξη, το Μάρτιο περίπου. Οπότε θα λάβει χώρα μια υπουργική σύνοδος με τους Ινδούς στο Νέο Δελχή, ώστε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία. Um, Ποια είναι τα, ε, τα υπάρχοντα προβλήματα. Οι δασμοί για τα αυτοκίνητα, το θέμα των αλκοολούχων ποτών είναι ακόμα υποσυζήτηση ε, και υπάρχει το κεφάλαιο της βιωσιμότητας, η παιδική εργασία και, διάφορα άλλα θέματα. Η Ινδοί στην αρχή δεν ήθελαν ούτε καν να τα συζητήσουν αυτά λέγοντα ότι δεν έχει καμία σχέση με μια εμπορική συμφωνία, ξεπερνάει το πεδίο εφαρμογή μια εμπορική συμφωνία. Του καταστήσαμε σαφέ ότι έχει, έχει και παραέχει σχέση με μια εμπορική συμφωνία και ότι χρειάζεται ένα τέτοιο κεφάλαιο διότι μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει να προβλέπετε κάτι τέτοιο στις ε, εμπορικές συμφωνίες, επιμείναμε και τελικά συμφώνησαν να υπάρξει ένα κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα στην εμπορική συμφωνία που θα υπογραφεί με την Ινδία. Βεβαίως πρέπει να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση και εκεί θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, αλλά καταστήσαμε απόλυτα σαφές και έγινε αποδεκτό αυτό ότι θα υπάρξει ένα, ε, το σχετικό κεφάλαιο στην ε, συμφωνία. Αναφερθήκατε στην παιδική εργασία. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Πρέπει ε, να δούμε ο κάτι που συμβαίνει στη Γεωργία ή σε βιομηχανικό πλαίσιο. Πρέπει να ε, το δούμε προοδευτικά αυτό το θέμα, αλλά οπωσδήποτε θα καλυφθεί από τις συμφωνίες που θα υπογράψουμε. Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις σας και άλλοι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Ινδία πιθανώς να διατυπώσουν και εκείνοι ερωτήσεις. Ο Έντβαρ Κόσοσνίκ που ήταν ε, και η συγητή και στον οποίο αναφερθήκατε. Θα μιλήσω τσεχικά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τσεχικά. Κύριε Επίτροπε, εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην παρουσίασή σας τονίσατε το θέμα των ευρωπαϊκών προτύπων, διότι νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέσον για να προωθήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα από πλευράς ευρωπαϊκής νομοθεσίας και για να ανταποκριθούμε στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Εγώ είχα συντάξει και μία έκθεση επί του θέματος και ως εκπρόσωποι διάφορων πολιτικών ομάδων έχουμε συζητήσεις επί πολλών θεμάτων. Υπάρχει όμως ένα, μια κεντρική ιδέα όπου συμφωνούμε, δηλαδή για τη μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά τη μείωση της ε, γραφειοκρατίας και την αντιμετώπιση του διοικητικού άχθους έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προσυπογράφουμε όλοι και ολόκληρη η Επιτροπή ΙΜΚΟ συμμετέχει σε αυτή τη δικασία, όχι μόνο η συγγετής Κοζέσνικ. Και Όλες οι πολιτικές ομάδες και ιδιαίτερα ο Μάλκον Χάρμπορ, ο πρόεδρος, προώθησε την έκθεση αυτή για το μέλλον των ευρωπαϊκών προτύπων. Έχω μία ερώτηση να σας υποβάλω, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει πολύ σημαντική εργασία για να ορίσει να οριοθετήσει τη μελλοντική νομοθετική εργασία για τα πρότυπα, ως προς τα πρότυπα. Τι θα κάνουμε με το κεφάλαιο του συντονισμού. Νομίζω ότι η νομοθετική ατζέντα μας για το μέλλον και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτή την επιτομή ε, προτύπων ε, εσείς κύριε Ντεγούχτ, ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Μπαρνιέ θα ασχοληθούν αυτό το θέμα. Πώς θα συντονίσετε τις ε, προσπάθειές σας. Και τι κάνετε με τη ΣΕΝΕΛΕΚ και τα άλλα υπερεθνικά σώματα και φορείς. Πώς ε, συντονίζετε αυτή την έργαση. Θα ήθελα ο κύριος Ντεγκούχτ να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ίσως θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω, αλλά είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από το βαθμό συντονισμού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρίνω με τον συντονισμό μεταξύ εθνικών αρχών στα πλαίσια του Συμβουλίου και έχω κάποια άποψη επί του θέματος γιατί χρημάτισα υπουργός εξωτερικών υποθέσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και διαπιστώνει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα διαφορετικό ζώο, θα μπορούσα να πω. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική διοικητική δομή που αυτόματα οδηγεί σε στενή συνεργασία μεταξύ των ε, διαφόρων χαρτοφυλακίων. Βλέπουμε σε εβδομαδιαία βάση και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών, ότι υφίσταται αυτός ο συντονισμός. Στα πλαίσια της ΕΝΕΛΕΚ υπάρχει στενή συνεργασία Γι' αυτό δεν νομίζω ότι υφίσταται ένα ουσιώδες ζήτημα εδώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος ως προς το βαθμό συντονισμού, ενδοκινοτικού συντονισμού. Ωραία λέει ο Πρόεδρος, πολύ ενθαρρυντικό αυτό και από τη δική μας άποψη. Μιλάμε, θα μιλήσουμε για το έγγραφο της εμπορικής ανάπτυξης και των διεθνών σχέσεων, διότι είναι ζήτημα το οποίο, στο οποίο συμφωνήσαμε και ο συντονιστές Λούχιγκάρτ, ο πρώτος ομιλητής και όποιοι άλλοι θέλουν το λόγο. Κύριε Λούχιγκάρτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να θα μιλήσω στα αγγλικά αντί στα δανέζικα, διότι από όσο γνωρίζω ο Επίτροπος δεν κατέχει τόσο καλά τη δανέζικη γλώσσα, τη γλώσσα της ε, δανημαρκίας. Θα πρέπει να με συγχωρήσετε γιατί έφτασα κάπως καθυστερημένα και ίσως το θίξατε αυτό το ζήτημα. Η ερώτησή μου είναι απλή. Βλέπω εδώ στις σημειώσεις ότι θα αναβαθμίσετε τη σχέση με τους στρατηγικούς εταίρους, όπως είπα Κίνα και ούτω καθεξής. Θα φτάσουμε σε μία εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και ποια είναι η θέση της Επιτροπής ως προς την ε, μία ελεύθερη, μία εμπορική σχέση στα πλαίσια του ΠΟΕ. We have no δεν έχουμε σχέδια να διαπραγματευτούμε μια τέτοια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών δηλαδή. Αλλά έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ και προσπαθούμε να επιλύσουμε εκρεμή ζητήματα. Στις 16 και 17 θα έχουμε τον Διατλαντικό Οικονομικό Διάλογο στην Ουάσιγκτον. Έχουμε συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους ως προς την ε, ημερήσια διάταξη και νομίζω ότι θα έχουμε ε, ορισμένα άναντι αποτελέσματα έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ορισμένα πρότυπα και επίλυση ζητημάτων πριν φτάσουν τα προϊόντα στην αγορά. Και εργαζόμαστε επ' αυτού. Επίσης προσπαθούμε να ε, άρουμε ορισμένα ποσοτικά εμπόδια μη Α, μη δασμολογικά. Με συγχωρείτε. let me give you the example of chlorine chicken, for example. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε σχέση με ορισμένα προϊόντα, όπως ε, για παράδειγμα ως προς τα πουλερικά. Θα έχουμε ένα συνολικό σύστημα ελέγχου της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και στις ΕΠΑ μπορώ να σας πω εντάξει, μπορούμε τα πουλερικά να τα πλένουμε με χλωριούχα προϊόντα, με χλωρίνη. Γιατί δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό λένε στη ΣΥΠΑ. Αλλά προσπαθήσαμε εδώ και χρόνια να βρούμε κάποια λύση, δεν τη βρήκαμε και αυτό σχετίζεται με την ε, κατανόηση του κοινού, διότι οι νομοθέτες δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν εργάζονται καλώς ή είναι ισχυρογνώμονες και ούτω καθεξής. Έχει σημασία το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία ορισμένα ζητήματα ή ένα έθνος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με Τη είπα δεν είναι το δασμολόγιο, διότι οι δασμοί είναι πολύ χαμηλοί μεταξύ των δύο χωρών. Άρα το θέμα δεν είναι η μη τα μη δασμολογικά εμπόδια. Έχει συνταχθεί μια έκθεση, μάλλον ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αναφέρεται ότι Εάν μπορούσαμε να απομακρύνουμε τα μη δασμολογικά προσκόμματα μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίμιση δηλαδή, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν πιο ευεργετικά από το γύρο της Ντόχα. Το θέμα των μη δασμολογικών εμποδίων είναι κάτι το διαφορετικό. Είχαμε την νομοθεσία Jones, το αντιμετώπισε αυτό και στο Βέλγιο το νομοθέτημα Jones απαγορεύει την δραστηριότητα ε, πλοίων στις ΗΠΑ που ε, δεν μπορούν να ε, έχουν ακτοπλοϊκή δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο ανάγεται στο 1922. Στα πλαίσια αυτά, ο γύρος της Ντόχα μπορεί να σταθεί καθοριστικός. Μπορώ να πω ότι πλέον οι ΙΠΑ προσπαθούν να κλείσουν το γύρο της Δόχα. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, ε, απομένει να ειδωθεί. Θα το δούμε μέχρι τις επόμενες ε, καλοκαιρινές διακοπές. Θα δείτε ότι θα καταβληθούν ε, σοβαρές προσπάθειες από ΙΠΑ και άλλους εταίρους να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα. Η G5, η Βραζιλία, ε, η Ινδία, Κίνα και εμείς, η G5, δηλαδή η G5 συν 2, δηλαδή και η Ιαπωνία και η Αυστραλία, θα κληθούν στις Βρυξέλλες για να επανεκκινήσει ο γύρος της ε, Ντόχα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο άνοιγμα, μια μεγάλη ευκαιρία. Και έχει μεγάλη σημασία στην πολιτική αυτά τα ανοιχτά παράθυρα, δηλαδή οι νέες ευκαιρίες, γιατί πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός ως προς αυτά τα ανοίγματα και τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας θέσω και εγώ ορισμένες συναφείς ερωτήσεις ε, μετά από την απάντησή σας στον κύριο Λίκεγκάρντ. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα που ανακοινώσατε στην Ολομέλεια των Βρυξελών πριν από τρεις εβδομάδες νομίζω ότι προσπαθείτε να ευθυγραμμίσετε όλους τους στόχους του υπερατλαντικού διαλόγου ε, και να εξετάσετε περισσότερο τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, τα, τα και τα μακροπρόθεσμα πρότυπα για τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, για ε, τα έξυπνα προϊόντα, την νανομηχανική κλπ. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και με δικά μας ε, ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Μία από τις εξελίξεις που συζητήθηκαν έντονα όταν άρχισε ο διατλαντικός διάλογος ήταν το νομοθετικό πλαίσιο. Διότι πολλοί νομοθέτες σε εθνικά κοινοβούλια ή στην ε, Αμερικανική Βουλή, στο Κογκρέσο, ε, θα έφερναν ισχυρή αντίσταση σε αλλαγές που θα θέλαμε να εφαρμόσουμε. Παραδείγματο χάρη στο θέμα των σχέσεων με την Ιαπωνία. Τώρα όμως συμμετέχουμε έντονα σε αυτό το διάλογο και ήθελα να σας ρωτήσω εάν ε, πρέπει να δώσουμε στην κοινή μας προσπάθεια περισσότερη πολιτική ισχύ. Ο Επίτροπος ε, θα υπάρξει θα γίνει μια συνάντηση 6 με 8 Δεκεμβρίου για τον ε, διάλογο νομοθετικού περιεχομένου 6 με 8 Δεκεμβρίου στις Ηνωμένε Πολιτείε. Next meeting. 6 mm, με 10 στο Σαν Φρανσίσκο. 6 με 10 Δεκεμβρίου. Ωραία, οπότε εκεί θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία θα σας ενημερώσουμε μετά στις 16 και 17 Δεκεμβρίου. Οπότε αναμένουμε με ενδιαφέρον την, ε, τη συμβολή σας, τις παρατηρήσεις σας. Ας πούμε λοιπόν ότι ε, ο ασθενή περιού συζητούμε, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση υγείας μέχρι τώρα και είχαμε πολλές, είχαμε εις συζητήσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, για αυτά τα θέματα και οι δύο πλευρές και είπαμε ότι καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να αναρρώσει λίγο ασθενείς διότι αυτό είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και γι' αυτό αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και διαιρέσαμε σε δύο τμήματα τη συζήτηση. Από τη μία πλευρά τα θέματα στρατηγικής δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε κοινέ προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά και δεύτερον τα θέματα ε, που, ε, μελλοντικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αναφιόμενες τεχνολογίες η ανάπτυξη της ε, διατλαντικής αγοράς και και το θέμα των ε, προτύπων βεβαίως και της προτυποποίησης έτσι ώστε να εδραώσουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που αναφύονται προβλήματα ώστε να μπορούμε να προλάβουμε και να συντάξουμε, να προβλέψουμε τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις τα πρότυπα και η προσέγγιση σε νομοθετικά θέματα τα έχουμε συζητήσει ήδη στο ρυθμιστικό, στη Ρυθμιστική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου και θα πρέπει να τα συζητήσουμε ξανά μία μέρα πριν από την Ολομέλεια των διαφορετικών ε, φόρουμ που υπάρχουν μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν είπαμε θα τα συζητήσει 16 και με 17 Δεκεμβρίου και θα μας βοηθήσετε ελπίζω στην ατζέντα που θα συντάξουμε και σε ποια θέματα θέλετε. Το πρόβλημα των containers ε, ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα Θέματα λοιπόν για την ατζέντα. Έχουμε ήδη επισημάνει ορισμένα θέματα προτεραιότητος και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα και τέλος θέλουμε να επιτύχουμε και στενότερη συνεργασία στο διάλογο αυτών των υπερατλαντικών των νομοθετών. δεν μπορώ να είμαι ταυτόχρονα και στην Washington, αλλά πιστεύω ότι ε, την επόμενη φορά θα πρέπει να συνδυάσουμε τις ενέργειές μας ώστε να συμπίπτουν. Ο Πρόεδρος, πιστεύω ότι οι μέλη της Επιτροπής μας όντως ε, θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στη διαμόρφωση της, της διάταξης και στις παρατηρήσεις. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μία μακρά ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο άλλο θέλει να λάβει το λόγο πριν ολοκληρώσω. σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Είδατε πραγματικά το έντονο ενδιαφέρον από πλευρά τη Επιτροπή μα και πώ θα θέλουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί σα. Θα σας καλέσουμε λοιπόν και πάλι περίπου σε ένα χρόνο για να μας ενημερώσετε. Εν τω μεταξύ στο διάστημα αυτό θα παρακολουθούμε την ανάπτυξη των στρατηγικών που παρουσιάσατε και θα βοηθήσουμε στις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη του εμπορίου διεθνώς και προσβλέπουμε με ε, ικανοποίηση τη μελλοντική ε, έκδοση της έκθεσης για το διεθνές εμπόριο. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά θέματα και φακέλους στο γραφείο σας αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα με ικανοποιεί η πρωτοβουλία που λάβατε μέσα στα πλαίσια των G5 Thin, G5 plus. Ε, σας ε, εύχομαι λοιπόν ε, ε, κάθε επιτυχία πριν να αρχίσετε το νέο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ.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

Uh, Κυρίες και κύριοι, έχουμε καθυστερήσει λίγο, αλλά περιμένω να δω ότι είμαστε όλοι παρόντες, όσοι πρέπει να είμαστε παρόντες για την επόμενη συνεδρία, για να συζητήσουμε την πολύ σημαντική συζήτηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Προτού όμως το κάνουμε αυτό, θα καλωσορίσω ένα νέο μέλος της Επιτροπής, την κυρία Ερεγκοεν Πέρες. Καλωσορίσατε ορίσατε. Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε. Uh, so, uh, we're Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας για την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν έχουμε όλους τους σκιώδεις. Η κυρία Γκέπερτ, η κυρία Τούν δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα. Ούτε κάποιος άλλος, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα... Α, και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι επίσης εδώ. Μόλις μπήκε στην αίθουσα, τον καλωσορίζουμε. Δεν έχουμε αρχίσει, κύριε Τριανταφυλλίδη. Αρχίζουμε τώρα. Και ο κύριος Πέτρη νομίζω θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Έτσι δεν είναι. Και θα δούμε αν ο κύριος Έντεντχοφ από την Προεδρία είναι επίση παρόν. Πάντως, εάν ε, ε, δεν έχει αντιρρήσει ο εισηγητή, μπορούμε να αρχίσουμε λίγο πιο νωρίς. Άντρε Σβάμπ, με χαρά σου δίνουμε το λόγο για να μας πεις που έχουν φτάσει συζητήσεις, ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε και οτιδήποτε άλλο θέλεις να πεις ε, ως εισαγωγή προτού απαντήσουν οι σκιώδεις ε, και συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ο Σβάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους σχεώδης για το χρονοδιάγραμμα στην τελευταία μας συνεδρίαση όταν ο κύριος Τελιάνη ήρθε να μας δει δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να παρουσιάσουν τις τροπολογίες τους συνολικά 1600 ήταν οι τροπολογίες και είναι Λυπηρό που είναι τόσοι λίγοι οι συνάδελφοι παρόντες. Συμφωνώ, Πρόεδρε, ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο θέμα. Για ορισμένου συναδέλφου ίσω αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγκατέλειψαν την ιδέα να καταθέσουν τροπολογίες. 1600 τροπολογίες όπως σα είπα, τι εξέτασα όλε. Νομίζω ότι ε, τις, κατάλαβα όλες επίσης και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο έργο να τις λάβει κανείς όλες υπόψη. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα στο οποίο θέλουν να συμβάλλουν όλοι οι συνάδελφοι μέσα από τις τροπολογίες τους. Μετά την τελευταία ημερομηνία κατάστροπολογιών θα γίνει μια σύντηση με τους τυώδεις για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ε, οδηγία αυτή. Είχαμε κάποια προβλήματα αρχικά με τις μεταφράσεις στις διάφορες γλώσσες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, προχωρήσαμε πολύ και όλοι οι σκιώδεις ηγητές κατ' επανάληψη με διαβεβαίωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Γι' αυτό θεωρώ λογικό το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο να παρατείνουμε κάπως τη συζήτηση ώστε να μην γίνει η ψηφοφορία όπως είχε προβλεφθεί το Φεβρουάριο, δύο εβδομάδες αργότερα, δηλαδή το Μάρτιο. Οπότε θα έχουμε όλο τον Ιανουάριο στη διάθεσή μας για άλλες επαφές, Πρωτού, στις 26 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ψηφίσουμε για τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα έχουμε καταλήξει μέχρι τότε. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές που με βοήθησαν ιδιαίτερα να συντάξουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και έτσι μπορέσαμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμφωνούμε, οι διαβουλεύσεις αυτές θα γίνουν κάτω από τρεις οπτικές γωνίες. Πρώτον, να μην μειώσουμε το υπάρχον επίπεδο προστασίας καταναλωτών σε κανένα κράτος μέλος. τα 27 κράτη-μέλη και είναι δυνατόν να βεβαίως αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας. Δεύτερον, συζητήσαμε τον καθηγητή Μόντι τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου και το ζητήσαμε να ενοποιηθούν όλες οι προτάσεις και να εναρμονιστούν όλες οι προτάσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι το σημείο 2-3. Και γι' αυτό δεν θέλουμε βεβαίως να χάσουμε και την οπτική της εσωτερικής ε, αγοράς και να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη συζήτηση με μονομένων σημείων, όπως παραδείγματο χάρη στο κεφάλαιο 4, το άρθρο 22, που αναφέρει τις ε, νομικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν στην εσωτερική αγορά και αν μπορούμε αυτές να τις εναρμονίσουμε. Στη, προς το συμφέρον των καταναλωτών θα πρέπει αλλά και βάσει των προτάσεων του καθηγητή Μόντι, πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να καλύψουμε την πλευρά της παράδοσης προϊόντων ε, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές και προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη να καλύπτεται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο η όλη διαδικασία ε, παραγγελίας και παράδοσης. Ε, στην παράγραφο 2 του 22 υπάρχει ακόμα μία στάφια. Πώς θα μπορέσει ο καταναλωτής να ε, έχει επιλογή μέσων πληρωμής χωρίς να επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνες. Θέλουμε λοιπόν να έχει μία επιλογή στο πώς θα πληρώνει τις παραγγελίες του διότι συνήθως ναι μεν έχει μια επιλογή αλλά όλοι αυτοί οι τρόποι τον επιβαρύνουν περισσότερο με επιπλέον δαπάνες. Οι συμβιβαστικέ προτάσεις που υπάρχουν θα μπορέσω να τις συζητήσω όταν έχουμε ολοκληρώσει και όλες τις συζητήσεις με τους εσκιώδεις εισηγητές. Πάντως δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει το, την παράγραφο 22. Ε, θα συνεχίσουμε μετά τις διαβουλεύσεις με την παράγραφο 26. Ε, μέχρι τώρα στις, 27, στις 26, σε 26 κράτη μέλη, ενώ σε ένα κράτος μέλη, μέλος υπάρχει μία σάφια. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνο για τα εμπορεύματα από τη στιγμή που βρίσκονται στα χέρια του. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει εάν υπάρξει ζημία στο προϊόν από τη στιγμή που έχει παραδοθεί. Ποιος έχει την ευθύνη και από ποιο νομοθετικό πλαίσιο καλύπτεται όταν σημειωθεί μία... Ε, όταν το εμπόρευμα βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν στην οποία παραδόθηκε. Εδώ δεν έχουμε ακόμα διατυπώσει όλες μας τις προτάσεις και την συνυπευθυνότητα. Διότι από τη στιγμή που ο καταναλωτής έχει το προϊόν στα χέρια του, εάν υποστεί ζημιά από τη χρήση του προϊόντος θα μπορούσαμε ας πούμε να του δώσουμε μία προθεσμία δύο εβδομάδων να δοκιμάσει το προϊόν και αν υποστεί ζημία ή βλάβη από το προϊόν ή χαλάσει τότε να είναι υπεύθυνη η εταιρεία ή αυτός ο οποίος το παρέδωσε ή ο κατασκευαστής εκεί δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε συμφωνία. Το κεφάλαιο 4 είναι πάρα πολύ περίπλοκο, ιδίω όσον αφορά την ιεραρχία της χρήσης νομικών μέσων για τον καταναλωτή, ε, πώς δηλαδή μπορεί να υποβάλει ε, ζήτημα ε, ε, ε, πώς εφαρμόζεται το πλαίσιο εγγυήσεων των προϊόντων, τι εγγυήσει ισχύουν σε όλη τη διαδικασία από την παραγγελία στην παράδοση και στη χρήση. Όλα αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά περίπλοκα και πρέπει να καταλήξουμε σε λύση. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τα δικαιώματα εγγύησεων. Εδώ έχουμε διαπιστώσει ότι το, τα εθνικά δίκαια διαφέρουν πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Ε, προσπαθούμε και εδώ να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του, πλαισίου, του νομοθετικού πλαισίου εγγύσεων και αν μπορούμε να εναρμονίσουμε όλες αυτές τις ε, διατάξεις ε, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εδώ παρουσιάζονται πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Εγώ νομίζω ότι το θέμα των εγγύσεων ε, δεν θα μπορέσουμε να το εναρμονίσουμε και γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά τα σημεία να τα περάσουμε σημείο προς σημείο, γραμμή προς γραμμή με τους εισηγητές ε, διότι η συμφωνία σε αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Και περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι είχαμε ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο ε, που ήταν ένας ε, κατάλογος ψηφοφοριών που περιλαμβάνει όλες τις τροπολογίες που έχουμε και θα πρέπει να το ε, τηρήσουμε αυτό, αυτό το, το, σχολι, το σχολιασμένο κατάλογο τροπολογιών. Η κυρία Γκέπχαρτ, η οποία ενδεχομένω να θέλει να διαγράψει όλο το κεφάλαιο 4. Ε, της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Σβάμπ για την σύντομη εισήγηση που έκανε. Πράγματι, η τελευταία μας συνεδρίαση δεν κατέληξε σε εναρμόνιση, αλλά ήταν καρποφόρα και αποδοτική. Και νομίζω αυτός είναι και ο στόχος των εργασιών μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που προτείνεται να ψηφίσουμε αντί στις 9 ε, Δεκεμβρίου στις ε, einigen können. Ich glaube, es wäre keine gute Sache, wenn wir... στις 27 ε, Ιανουαρίου ε, διότι έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες επί των οποίων πρέπει να συμφωνήσουμε. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν όλα αυτά να τα κάνουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα σε ένα σημείο. Άκουσα ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ή εσείς θέλετε να προτείνετε τη σύνταξη μιας μελέτης για την αξιολόγηση της συμπερίληψης ψηφιακών προϊόντων. Δηλαδή τι θα γίνει αν συμπεριληφθούν ε, και τα ψηφιακά προϊόντα. Ε, θα μπορέσουμε να το καλύψουμε αυτό και μέσα στα πλαίσια του συμβασμού. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να συμπεριλάβουμε και τα ψηφιακά προϊόντα και θα ήθελα να με ενημερώσετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της προφορικής ερώτησης. Για το άρθρο 20 δεν έχουμε βρει ακόμα συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν ορισμένα εκρεμή ε, ζητήματα και περιμένω πραγματικά με ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, ιδίως όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης, διότι εκεί έχουμε ακόμα ορισμένα σημεία ασαφή πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα της παράδοσης ε, προϊόντων. Ιδίως όταν ένας, ε, μια επιχείρηση, ένας ε, έμπορος εγγυάται ή λέει ότι θα παραδώσει το προϊόν μέσα σε 48 ώρες και δεν μπορέσει να σεβαστεί αυτή την προθυσμία, πιστεύω ότι είναι αδιανόητο να μην του δώσουμε μια άλλη ευκαιρία πέραν των 48 ώρων. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια ε, ζητήματα τα οποία ακόμα εξετάζουμε και που δεν έχουν συμφωνηθεί. Το άλλο σημείο που θίξατε, το πώς θα πληρώνει ο καταναλωτής, ε, με τι μέσα πληρωμών υπάρχουν και ε, δεδομένου ότι πολλές φορές εμπλέκονται επιπλέον δαπάνες τον τρόπο πληρωμής πρέπει να το συζητήσουμε λεπτομερώς διότι δεν φτάνει να πούμε ότι θα βρούμε ένα νέο τρόπο ή ένα άλλο μέσο πληρωμής. Ε, Παραδείγματο χάρη στη Γερμανία έχουμε μια αεροπορική εταιρεία που όταν πλήρωνες έλεγε ότι δεν θα επιβαρυνθείς ε, περισσότερο άμα πληρώσεις με αυτόν τον τρόπο μέσω αυτού του συστήματος αλλά πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι ήξεραν ή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αδάπανο σύστημα λοιπόν ε, τιμωρήθηκε πήγε στο δικαστήριο και της επευλήσει ποινή. Δεν, είναι λοιπόν ε, εύλογο να πούμε ότι οι πληρωμές θα γίνονται μέσω του συστήματος ε, ΩΜΕΓΑ όταν οι άνθρωποι δεν έχουν, οι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα αυτό παρόλο που είναι αδάπανο, δεν επιφέρει επιπλέον δαπάνες. Ε, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας, όπου διαφέρουν οι απόψεις μας και Όσον αφορά το κεφάλαιο 4, είπατε ότι μάλλον δεν μπορείτε να προβλέψετε μία εναρμόνιση, πλήρη εναρμόνιση. Τουλάχιστον αν δεν επιτύχουμε εναρμόνιση, θα αφήσουμε περιθώρια ευελιξίας στο κεφάλαιο 4. Π.χ. δεν μπορούμε να ορίσουμε ντε και σόνι ότι ο τρόπος πληρωμής σε παραγγελίες, σε εμπορικές συναλλαγές online θα είναι μόνο οι πιστοτικές κάρτες. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία ευελιξία μια ευελιξία για τον καταναλωτή, τι, μέσο πληρωμής θα επιλέξει και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ορίσουμε τελικά εσφαλμένες, να μην διαλέξουμε εσφαλμένες διαδικασίες που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και θα δυσκολέψουν τον καταναλωτή στις συναλλαγές του. Ευχαριστώ. Okay, well, I think, um, Νομίζω και συμφωνώ με την κυρία Γκέπχαρτ στο θέμα του χρονοδιαγράμματος Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα στο έπακρο ε, σε σχέση ιδιαίτερα και με τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που ήθελε ο εισηγητής να συζητήσουμε και το συζητήσουμε και στο, στους συντονιστές. Ο κύριος Ροσφόρ και μετά ο κύριος ε, Τριανταφυλλίδης στη συνέχεια. Ο κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Σβάμπ για την ε, πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε έχοντας να, αντιμετωπίσω, να αντιμετωπίσει 1600 τροπολογίες οι οποίες σχεδόν έχει μάθει απ' έξω. Θα το δούμε αυτό εάν υποβάλουμε γραπτή ερώτηση. Η αναβολή της ε, τελικής ημερομηνία για την κατάσταση των τροπολογιών είναι μια καλή και μια δυσάρεστη είδηση. Καλή είδηση, δεν χρειαζόμαστε χρόνο για να δουλέψουμε αποτελεσματικά. Δυσάρεστη είδηση ότι επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για πολύ δύσκολο εγχείρημα και δεν έχουμε ακόμα βρει όλες τις λύσεις. Μου λένε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι απέσυρε από τη συνεδρίαση της 10 η Δεκεμβρίου ε, το Συμβούλιο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό αλλά υπάρχουν φαίνεται δυσκολίες από παντού. Ας μην κρυβόμαστε, μην, κρυβ, μην ε, ε, αρνιόμαστε να δεχθούμε την αλήθεια. Αυτό είναι ένα δύσκολο κείμενο. Έκανα, είχα μια εμπειρία πριν από την τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο και παρόλο που είμαι κάποιος που γνωρίζει καλά το κείμενο προσπάθησα να το ξαναδιαβάσω σαν να ε, το έβλεπα. και δεν είδα μια κατευθυντήρια γραμμή και είναι δυσάρεστο όταν δεν βλέπουμε μια κατευθυντήρια γραμμή σε ένα κείμενο, όταν έχουμε την αίσθηση ότι δεν ε, καλύπτονται όλες τις λεπτομέρειες, αυτό σημαίνει ότι η δουλειά δεν έγινε σωστά. Το λέω διότι αυτό έχω το αίσθημα, αυτό ήταν το αίσθημα που ένιωσα όταν διάβασα αυτό το κείμενο. Ο Ανδρέας δικαίως ε, είπε ότι δεν θέλουμε να, να οπισθοδρομήσουμε σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Αυτή η οδηγία δεν φτάνει κάποια στιγμή. Αλλά φτάνει τη στιγμή που οι πολίτες και οι καταναλωτές έχουν πια κουραστεί και έχουν δισταγμούς για την εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα μιλάμε για την κατανάλωση. Το πιο Η πιο καθημερινή δραστηριότητά τους ε, και στις σχέσεις τους με την ενιαία αγορά, με την ιστορική αγορά, έστω και να τη χαρακτηρίζουν έτσι. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Το κείμενο αυτό να, ε, να ρίξει φως σε ορισμένους τομείς επιτρέποντας καταναλωτές να έχουν λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη ότι θα τους προσφέρει περισσότερα προϊόντα με καλύτερες νομικές ε, προϋποθέσεις και με καλύτερες τιμές η ενιαία αγορά αλλά υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσει ο καταναλωτής ένα κείμενο που τον απομακρύνει από την Ευρώπη και του δίνει την εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζει σωστά τα πράγματα η Ευρώπη και αυτό θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που οι αρχέ των κρατών μελών θα το πουλήσουν αυτό το κείμενο κατά την ενσωμάτωσή του στην εθνική του νομοθεσία. Θα λένε απλώ ότι πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα γιατί μα το επιβάλλουν οι Βρυξέλλε οδηγώντα σε εσωτερικέ διαμάχε και ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των καταναλωτών, έστω και αν δεν ισχύει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει η οδηγία, αλλά θέλω να δω τι θα συμβεί μετά την έγκρισή τη Εφόσον μιλάμε για μια οδηγία ε, που αφορά την κατανάλωση, αυτό είναι σημαντικό, να δούμε τι θα γίνει κατά την εφαρμογή της. Στις συναντήσεις που θα έχουμε, πρέπει να αναζητήσουμε σαφήνεια, απλούστευση, να αποφύγουμε οτιδήποτε που θα είχε ως αποτέλεσμα, θέλω να το ξαναπώ, μπορεί να ακούγεται σαν ευσεβής πόθος, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν, ε, την, σαν ε, την, ε, η αναζήτηση κάποιου ε, κάποια ιδεώδους κατάστασης αλλά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για συμβιβασμό για αυτό το κείμενο αν επρόκειτο να το ψηφίσουμε με μια ομάδα που το υποστηρίζει και μια ομάδα που δεν το υποστηρίζει πρέπει να γίνει να βρούμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά στον καταναλωτή στην ενιαία αγορά. Γι' αυτό χρειάζεται να αναζητηθεί ένα συμβιβασμό. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Και κάτι που δεν είπε ο Ανδρέας. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά η πρόταση αλλαγή του χρονοδιαγράμματο προέκυψε από τη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών τη περασμένη εβδομάδα, παρόλο που υπήρχαν και άλλοι λόγοι, αλλά σε αυτή τη συνάντηση αφιερώσαμε σχεδόν δύο ώρες εξετάζοντας 1,5 άρθρο και δεν καταλήξαμε οριστικά. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Το άρθρο 22 είναι ένα άρθρο που καλύπτει πολλά άλλα, εμπεριέχει πολλά άλλα αλλά δείχνει, δείχνει πόσο ευρύ είναι το θέμα αυτό το παράδειγμα. Από πολιτική άποψη θα ήθελα τώρα να πω και αυτή είναι η άποψη της ομάδας μου. Ε, έχουμε δύο πολιτικές προτεραιότητες σχετικά με αυτή την οδηγία. Η πρώτη είναι ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αν υπάρξει κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι οι πωλήσει από απόσταση προτιμούμε μία οδηγία που να εστιάζεται σε αυτό το θέμα των πολυλήσεων από απόσταση παρά να πάρουμε μία οδηγία που να προσπαθήσει, προσπαθεί να καλύψει τα πάντα χωρίς να προσφέρει κανένα νέο στοιχείο. Και όσο περισσότερο επιμένουμε να θέλουμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές κατανάλωσης, τόσο περισσότερο διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην εστιαστούμε στα σημαντικά θέματα, χρησιμοποιώντας γενικές διατυπώσεις που δίθεν εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά τα δικαιώματα καλύπτονται και προστατεύονται απόλυτα. Και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου, εφόσον ε, μιλήσαμε για το κεφάλαιο 4 υπάρχουν πράγματι σε αυτό το κεφάλαιο πολλά πράγματα που προτείνονται που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα καλύψουμε όλα ας σκεφτούμε λοιπόν πως θα, αποφύγουμε από το να ξεχάσουμε το βασικό στόχο, το βασικό σκοπό. Όπως είπε ο Άντρε Φουάμπ ε, πρέπει να ξαναδούμε το άρθρο 22, το θέμα των παραδόσεων, το θέμα των ε, συστημάτων πληρωμής. Ο Ανδρέα Σουάμπ ανέφερθηκε ναι, στην ιεράρχηση των ε, ένδικων μέτρων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δικαιωμάτων καταναλωτών που πρέπει να πλουστεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα που θα ιεραρχεί τα ένδικα μέσα με διάφορους τρόπους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν, να επιλέξουν ή όχι καταναλωτές είναι κάτι που μπορεί να οδηγεί σε στρεβλώσεις και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε για τις μεθόδους πληρωμής η κυρία Γκέμπερτ. Είναι σαφές και πρέπει να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα και θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον εισηγητή. Όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένας τρόπος πληρωμής που να είναι, ένας τρόπος πληρωμής που να είναι δωρεάν, αυτό σημαίνει ότι γίνεται αυτό για να διευκολύνουμε τις ε, πωλήσει από απόσταση. Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε τις πωλήσει μέσω ίντερνετ και από απόσταση αυτό δεν τις διευκολύνει. Όπως είπε η κυρία Γκέμπερτ πρέπει να είναι ένα καθιερωμένο ε, τρέχον σύστημα ε, πληρωμών αλλά και σύγχρονο και εξυγχρονισμένο σύστημα πληρωμών. Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η επιχείρηση που λέει σας υπόσχομαι μία παράδοση σε μία δεδομένη προθεσμία στα πλαίσια της πολιτικής του marketing πρέπει να θεωρηθεί ε, ότι είναι μια υπεύθυνη επιχείρηση. Αλλά πρέπει να δούμε και τη σημερινή πραγματικότητα. Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, μιλάμε για παραδόσεις που δεν γίνονται τις ημερομηνίε μέσα στις προθεσμίες που είχε ε, ανακοινώσει η εταιρεία διότι μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα στην παραγωγή, στον εφοδιασμό κτλ. Πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και να καλύψουμε και αυτό το θέμα στην οδηγία. Γι' αυτό ε, ε, υπέβαλα τροπολογίες και όπως είπε η κυρία Γκέμπαρτ, αν μια επιχείρηση πει θα παραδώσει 48 ώρες, αν δεν παραδώσει 48 ώρες, προτού ο καταναλωτής μπορέσει να ακυρώσει ε, το, την αγορά του η επιχείρηση μπορεί να θεωρήσει ότι έχει καθυστερήσει, ευθύνεται γι' αυτό. Εάν δεν όμως παραδώσει χωρίς να ξεπεραστούν οι 48 ώρες, δεν ε, μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση εκτός Πρόκειται για πάρα πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες ε, αναφέραμε. Αν πρόκειται για παράδοση ε, μια τουρτα γενεθλίων και φτάσει η τούρτα δύο μέρες μετά τα γενέθλια, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν με ρεαλισμό συμβιβαστικές λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις οικονομικές συνθήκες, χωρίς παραχωρήσεις προς τα δικαιώματα. Υπάρχουν πολλά δικαιώματα που δεν είναι γνωστά από τους καταναλωτές, παρόλο που είναι δικαιώματα που τους αφορούν. Και αν δεν ε, τα προσδιορίσουμε αυτά, δεν θα, είμαστε, δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει με δίκιο και σωστό τρόπο τους καταναλωτές. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και η παράταση των προθεσμιών θα μας βοηθήσει να, εργαστούμε, να συνεργαστούμε και να αναζητήσουμε συμβαστικές λύσεις. Uh, ευχαριστώ κύριε Ροσφόρ που προσπαθήσατε ε, με, επιτυχία θα έλεγα να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε συγκεκριμένα σημεία της ε, πρότασης γιατί θέλουμε ε, ουσιαστικά να προσφέρουμε μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές μας. Και έτσι θέλουμε να ερμηνευθεί η οδηγία ότι και τους καταναλωτές βοηθά και προστατεύει αλλά και την εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια περιφερειακή ισορροπία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να επιτύχουμε πρόοδο και να βελτιώσουμε ο κύριος Τριανταφυλλίδης παρακαλώ είναι ο τελευταίος σκιώδης εισηγητής και ο κύριος Κόζιτσικ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε με τον εισηγητή οι σκιοδησηγητές, παρόλο που υπάρχουν τόσο διαφορετικές απόψεις, καταφέρουμε να επιτύχουμε πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα που αναβλήθηκε μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, όπως πρότεινε ο κύριος Σβάμπ, για να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για τις ε, απαραίτητες συζητήσεις. Είναι απολύτως αναγκαίο να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Ε, γι' αυτό ε, συμφωνώ απόλυτα με την αναβολή για τις 27 πρώτου. Ωραία. Έχουμε και άλλους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες, ο κύριος Λαχνά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ υπέβαλα αρκετές τροπολογίες και συμφωνώ με τον κύριο Ροσφόρ, ο οποίος συμφώνησε με την κυρία Γκέπαρτ. 1600 τροπολογίες πρέπει να τις χειριστούν οι σκιώδεις εισηγητές. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω αυτό το έργο. Θα ήθελα όμως ε, να ψηφίσω κι εγώ ε, ευσυνείδητα. Όταν ε, μιλήσετε με νομικούς εμπειρογνώμονες, μας λένε πώς είναι δυνατόν να διαβουλεύετε το κοινοβούλιο και να θεωρείτε σοβαρό σώμα όταν έχει αυτό το, τον όγκο, τη χιονοστιβάδα των τροπολογιών έχετε δίκιο λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε ε, μεν το φιλόδοξο πρόγραμμα της ε, πρότασης ε, της Κομισιόν αλλά πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτό το, το μνημειώδες έργο. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μας απασχολούν με πάρα πολλές παραμέτρους και πρέπει όλες αυτές να τις συζητήσουμε. Εγώ ως Ευρωβουλευτής λέω ε, αν ο εισηγητής συμφωνήσει με τους κοιόδης εισηγητές, τι θα γίνει στην τελική ψηφοφορία, τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Ο καθένας θα έχει ελεύθερη ψήφο. Ε, πώς λοιπόν θα γίνει όλη η διαχείριση αυτού του θέματος. Αυτό το οποίο ε, έχουμε φορτωθεί τώρα είναι ένα διοικητικό χάος μία τερατώδης κατάσταση η οποία έχει αναπτυχθεί ε, διότι αυτά τα οποία έχει προτείνει η Κομισιόν δεν είναι ε, ριζοσπαστικές ή επαναστατικές αλλαγές της κατεύθυνσης γενικά της ε, εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών. Όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς περιορίζεται θα έλεγα σε δύο σημαντικά θέματα. Καταρχάς, οι εμπορικές συναλλαγές εξ αποστάσεως. Επίσης, διευρύνεται λοιπόν ο ορισμός των συναλλαγών εξ αποστάσεως. Επίσης, ε, ε, ευρύνονται, ευρύνονται ερμηνευτικά άλλες, ε, άλλοι ορισμού και η Κομισιόν δεν μας εξηγεί γιατί αλλάζει τους ορισμούς και πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Εάν λοιπόν δεχτούμε τις προτάσεις της Κομισιόν επειδή δεν μπορούμε να χειριστούμε σε βάθος 1600 τροπολογίες κινδυνεύουμε να περάσει κάτι το οποίο θα επηρεάσει δυσμενώς τους, τους, τους εμπορευόμενους και τους καταναλωτές. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρές οικογενειακές ε, μονάδες από έναν-δύο οι οποίοι πουλάνε αγαθά ε, στο διαδίκτυο και όλοι αυτοί οι ελάχιστες μικρομονάδες θα επηρεαστούν από όλον αυτό τον όγκο των αποφάσεων ε, δεν πρόκειται εδώ μόνο για μεγάλες εταιρείες αλλά πρόκειται και για πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί κάποιος ε, συνταξιούχος παραδείγματο χάρη να ασχοληθεί με όλο το νομοθετικό πλαίσιο της ε, προστασίας των καταναλωτών και να μελετήσει όλες τις νομοθετικές επιπτώσεις των 1600 τροπολογιών. Εγώ δεν είμαι συνταξιούχος, ούτε συνταξιούχος δάσκαλος και δεν έχω ούτε τις γνώσεις ούτε τον καιρό ε, να το κάνω αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει το κεφάλαιο 5 να διαγραφεί πλήρως γιατί δεν χρειάζεται, δεν είναι αναγκαίο δεν πιστεύω ότι όλο το δίκτυο προστασίας καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να καταρρεύσει. Δεν βλέπω δηλαδή καμία τεράστια καταστροφή μπροστά μας. Ε, να διατηρήσουμε τα κεφάλαια 1, 2, 3. Πιστεύω ότι είναι λογικό το περιεχόμενό τους. Προσφέρει την, την ελάχιστη προστασία, τις ελάχιστες διατάξεις. Δηλαδή το αναγκαίο κατόφλι παρέμβασης και ρύθμισης και νομίζω ότι τα άλλα όλα είναι περιτά. Βεβαίως υπάρχουν τροπολογίες και πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι επίγον αυτό το θέμα ε, διότι εμένα με ενδιαφέρει, είναι λίγο προσωπικά αυτά τα θέματα, αλλά ε, σαφώς υπάρχουν και τομείς που χρειάζονται περισσότερη προστασία, αλλά δεν μπορούμε όλα αυτά να τα χειριστούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που αποφάσισε το Κοινοβούλιο στην Πράσινη Βίβλο, αυτά πρέπει να ισχύουν. Απλούστευση, απλοποίηση, εντάξει, ε, συμφωνία στα ελάχιστα πρότυπα, ε, τα τέσσερα και πέντε κεφάλαια να διαγραφούν, να διατηρήσουμε τα κεφάλαια 1, 2, 3 και να τελειώνει η ιστορία, διότι μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, έκανε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Αλλά αυτό που κάνουμε συνεχώς είναι να διασπάμε σε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Παίρνουμε δηλαδή μία, ένα νομοθετικό μέσον και το κατατεμαχίζουμε σε χίλια κομμάτια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ενσωματώσουμε, να εναρμονίσουμε στο ελάχιστο επίπεδο, αλλά να μην επισέλθουμε ε, κατευθείαν σε, σε μια τέτοια τεράστια πρόταση που να πρέπει να ψηφίσουμε. Ας προχωρήσουμε βήμα προς βήμα και πιο αργά. Προστείνω λοιπόν να διαγραφεί όπως είπα το ένα μέρος της πρότασης 4-5 και να διατηρήσουμε το κεφάλαιο 1-2-3 και να χειριστούμε έτσι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την ξεκάθαρη θέση σας και μπορεί να υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις από τα μέλη μας. Εν τω μεταξύ έχω τον κύριο Χουανόχο και την κυρία Βάιλερ. Ο κύριος Χουανόχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ αρχής η πολιτική μου ομάδα και εγώ βεβαίως είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την πλήρη εναρμόνιση που επιθυμεί η Κομισιόν. Είμαι ευγνώμων στον κύριο Σβάμπ διότι προσπάθησε να βρει μια ενδιάμεση οδό μεταξύ της πλήρους εναρμόνισης και της ελάχιστης εναρμόνισης. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, όμως υπάρχουν ανεπάρκειες ως προς ε, ενδεχόμενες εγγύησεις προς τον καταναλωτή. Και το οικοδόμημα είναι σαθρό και από νομικής πλευράς. Επί της ε, ουσίας νομίζω ότι ο κύριος Σφάπ κάνει το ίδιο λάθος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η μέγιστη εναρμόνιση είναι το σημείο εκκίνησης. Ενώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε σημείο προς σημείο πώς μπορούμε να ε, υπερασπιστούμε τον καταναλωτή πριν φτάσουμε στην πλήρη εναρμόνιση. Έχω υποβάλει γύρω στις 30 τροπολογίες έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή ως προς, τα, ε, ως προς την πληροφόρηση και την καταγγελία μιας ε, συμφωνίας. Επίσης θα πρέπει οι πληροφορίες προς τον καταναλωτή να βοηθούν τον ίδιο τον καταναλωτή να έρχεται σε επαφή με τους παρασκευαστές. Δυστυχώς όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο μέσω διαδικτύου και μια ταχυδρομική διεύθυνση δεν αρκεί ως σημείο επαφής. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει μια απλή ε, προφορική συμφωνία τηλεφωνικός γιατί τα θύματα είναι οι καταναλωτές και μόνο με την υπογραφή της, ε, του συμβολέου ε, αναλαμβάνει ευθύνες ο καταναλωτής. Ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης, νομίζω ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης των 14 ημερών από την ημερομηνία ε, συμφωνίας θα πρέπει να ισχύει. Ως προς την πώληση αγαθών τότε οι 14 μέρες αρχίσουν να μετρούν από τη στιγμή που θα παραδοθεί το προϊόν. Επίσης θα πρέπει να οριστεί μία προθεσμία 30 ημερών, διότι πολλές φορές ε, αρχίζει κανείς να αγοράζει ας πούμε έπιπλα ένα μήνα πριν από τη μετακόμιση και τότε συμφωνείται μεταξύ ε, κατασκευαστή και καταναλωτή καταναλωτή η ημερομηνία παράδοσης. Γι' αυτό θα πρέπει τα συμβαλόμενα μέρη να ε, μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους ευθύνες και μέσα στα πλαίσια του δικαιώματος υπαναχώρησης. Αν κάποιος αγοράσει έναν τεράστιο καναπέ, όταν παραδοθεί ο καταναλωτής δεν θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα ε, η τη στιγμή που θα πρέπει να πληρώσει τη μεταφορά. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να υπομειστεί το κόστος ε, επαναπαστολής ε, του αγαθού τη στιγμή που υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Επίσης, ο, ο καταναλωτής θα πρέπει να αποφασίσει ως προς ε, το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα ενός ελαττωματικού προϊόντος, δηλαδή τι θα γίνει σε αυτή την ε, περίπτωση. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βανλόκ. Η κυρία Βάιλερ. <clears throat> Ευχαριστώ. Είχα ζητήσει το λόγο όταν άκουσα τη φουριόζικη παρέμβαση του κυρίου Λέχνερ, την ενθουσιώδη, παθιασμένη θα έλεγα, ε, και θέλει να απορρίψουμε σχεδόν το μισό ντοσιέ. Και να ξαναρχίσουμε αυτού και από την αρχή μετά από δύο-τρία χρόνια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν και οι πολιτικές ομάδες τη θέση τους. Τώρα, δεδομένου θα ψηφίσουμε αύριο την ε, μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων, πιστεύω ότι εδώ διακυβεύονται ορισμένα συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, Ορισμένες τροπολογίες που αφορούν μελέτες επιπτώσεων είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Άρα όταν ψηφίσουμε αύριο στις 10 θα πρέπει οι συντονιστές να συμφωνήσουν και να πούμε ότι η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο θεωρεί πολύ σημαντικό να γίνει μια νέα μελέτη αξιολόγηση επιπτώσεων σε αυτό το πακέτο των τροπολογιών. Ε, το αφήνω αυτό στα χέρια των ικανών ε, εισηγητών, αλλά θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε αυτή τη δυνατότητα της μελέτης, αξιολόγησης επιπτώσεων. Ε, διότι ίσως προκύψει κάτι που δεν το, πρόλα... δεν το πρόβλεψε κανείς μας. Νομίζω ότι αυτό συμβαδίζει με την αυριανή ψηφοφορία σε σχέση με μελέτες αντικτύπου. Υπάρχει και ένα επιπρόσθετο έγγραφο στις ε, τροπολογίες FAB και θα πρέπει να υπάρχει μία ε, μελέτη αντικτύπου σε στις 1.300 ε, τροπολογίες. Σε σχέση όμως με τα ψηφιακά προϊόντα, 1.600 τροπολογίες, με συγχωρείτε, θα πρέπει να δούμε εκ του σύνεγγυς όλα αυτά τα δεδομένα για να δούμε πώς αναλαμβάνει η Επιτροπή αυτό το έργο. Και θα θέλαμε ο κύριος Πέτρη να απαντήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν νομίζω ότι είχε εκφράσει τις απόψεις του σε σχέση με τα ψηφιακά προϊόντα και τις σχετικές τροπολογίες. Επίσης, στα ζητήματα Λέχνερ σε σχέση με τα πρόσθετα κεφάλαια, Νομίζω ότι και το Συμβούλιο εξετάζει αυτό το θέμα και θα ήθελα να μάθω τι θα μας πει ο κύριος Πέτρη. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να συνεισφέρουν στη συζήτηση κατά πόσο ο εισηγητής ε, θέλει να πει κάτι. Να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και μετά θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Πέτρε από την Κομισιόν να μας μιλήσετε για όσα ακούσατε μέχρι τώρα και αν υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφού άκουσαμε με ενδιαφέρον τις σημερινές συζητήσεις, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω αυτή τη διαδικασία προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ θετικό το ότι βρήκατε το χρόνο για να διερευνήσετε τις διάφορους, διάφορες οδούς για να μπορέσετε να φτάσετε σε ένα συμβιβασμό μέσα στον Ιανουάριο. Εντάχει, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα ως προς τα σχόλια, ορισμένα εξειδικευμένα σχόλια ως προς την παράδοση. Το θέμα της παράδοσης εθίγει από διάφορα μέλη και συζητήθηκε και στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορώ να σας πω, ο κύριος Ροσφόρ αναφέρθηκε σε αλλαγές έτσι ώστε να μην υπάρξει άμεση πάυση του συμβολέου τη στιγμή που ο καταναλωτής θέλει το προϊόν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Εδώ γίνονται και συζητήσεις στο Συμβούλιο που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Ε, η, το θέμα της απόστασης και των πωλήσεων εκτός καταστήματος η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να διευρύνει την εμβέλεια της οδηγίας σε σχέση με τις ε, τηλεπολίσεις ή τις πωλήσει εκτός καταστημάτων. Θέλουμε να, αυξήσουμε την, να επαυξήσουμε την προστασία του καταναλωτή και να κλείσουμε τα κενά που υπάρχουν στην ε, παρούσα οδηγία, έτσι ώστε οι καταναλωτές σε εξαποστάσεως συμβάσεις να μην πρέπει να γνωρίζουν ε, επακριβώς όλες ε, τις ρήτρες μιας τέτοιας σύμβασης τη στιγμή που έχει ζητηθεί τουλάχιστον η επίσκεψη του εμπόρου σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και για να κλείσουμε κενά τα οποία δημιουργήσαν ε, προβλήματα στους καταναλωτές. Ο κύριος Χουαγνόκ αναφέρθηκε στις προφορικές συμβάσεις, σύναψη προφορικών συμβάσεων που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν γραπτός. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο και θα ήθελα να λάβετε υπόψη <coughs> ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επαχθές για το τηλεμάρκετινγκ. Τη στιγμή που χρειάζεται πάντα επαναεπιβεβαίωση αυτών των συμβάσεων γραπτός. ως προς τη μη καταβολή πληρωμών κατά την περίοδο υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης. Αυτό είναι επαχθές για τον έμπορο, κατά την άποψη της Κομισιόν. Και όταν μιλάμε για ογκώδη αγαθά, το θέμα αυτό μπορεί να επιληθεί διαφορετικά. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής να μην αναλάβει το κόστος επαναποστολής. Να υπάρχει ένα όριο, ας πούμε. Ο καταναλωτής να μην καταβάλει το κόστος πάνω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Ή να έχουμε ειδικού κανόνες για ογκώδια αγαθά, όπως συζητήθηκε και στο Συμβούλιο. Τέλος, Πρόεδρε, ως προς το θέμα των ψηφιακών ε, αγαθών που θίξατε. Η Επιτροπή δεν έχει εισαγάγει κανόνες για το κατά πόσο ε, συμβαδίζουν, συμφωνούν, μάλλον συμμορφούνται αυτά τα προϊόντα ως προς τον κανονισμό Πιστεύουμε ότι τα ψηφιακά προϊόντα καλύπτονται από τις άλλες πτυχές της ε, ε, πρότασης, δηλαδή στα κεφάλαια 3 και 5, τηλεμάρκετινγκ και εκτός καταστήματος πωλήσει. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν και για τα ψηφιακά αγαθά, όπως είχε σχεδιαστεί. Ως προς το θέμα της συμμόρφωσης που ε, θίγει στα πλαίσια της ε, Πράσινης Βίβλου έγινε μία διαβούλευση οι ενώσεις καταναλωτών θέλαν να υπάρχουν κανόνες δυνάμει του κεφαλαίου 4, ενώ οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας έθιξαν πληθώρα προβλημάτων σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο πλήττονται οι καταναλωτές τη στιγμή που είναι ελαττωματικά τα ψηφιακά προϊόντα και που χρειάζεται, όπου χρειάζεται ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο. Γι' αυτό θα μελετήσουμε το ζήτημα εις βάθος και έχουμε δύο μελέτες Η μία θα ασχοληθεί με την οικονομική πτυχή του θέματος. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγια προς τους καταναλωτές και οι καταναλωτές θα ορίσουν τα προβλήματα και θα, τα, θα, θα, θα δουν κατά πόσο υπάρχουν ε, απτές ζημίες προς τον καταναλωτή δηλαδή, κατά του καταναλωτή. Έτσι ώστε να είναι ε, μετρήσιμες οι επιβλαβείς επιπτώσεις. Η άλλη πλευρά της μελέτης ασχολείται με την νομική πλευρά του ζητήματος, δηλαδή πώς ρυθμίζονται αυτά τα προϊόντα από τα κράτη-μέλη, από τις εθνικές νομοθεσίες και ποια συμπεράσματα συνάγουμε από αυτό. Πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα της συμμόρφωσης των ψηφιακών προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ε, διενεργούνται οι μελέτες. Δεν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συμπεράσματα. Έχουμε λάβει ορισμένες πληροφορίες για την νομική κατάσταση στα κράτη-μέλη που είναι ιδιαίτερα σαφής και αποκλίνουσα και θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011. Ίσως ε, είναι δύσκολο να γίνει χρήση αυτών των ε, αποτελεσμάτων στην ε, παρούσα διαπραγμάτευση στο παρόν στάδιο της ε, διαπραγμάτευσης. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα των ε, μελετών ή της δαυτής, διτής αυτής μελέτης θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα χειριστούμε τα ψηφιακά προϊόντα σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Από ό,τι μας είπατε αντιλαμβάνομαι ότι η της δαυτης διτης αυτης μελετης θα δουμε πως θα αντιμετωπισουμε πως θα χειριστουμε τα ψηφιακα προιοντα σε ενα συγκεκριμενο νομοθετικο πλαισιο ευχαριστω απο οτι μου ειπατε αντιλαμβανομαι οτι η επιτροπη δεν συμφωνεί με τις τρεπολογίες. Μπορεί να μην το είπατε έτσι ευθέως. Μας είπατε ότι προτιμάτε να περιμένετε μέχρι τα μέσα του 2011 που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναδούμε γύρω από τα τέλη του επόμενου έτους αυτή την οδηγία. Πάντως πρέπει να δούμε τι πιστεύουν οι συνάδελφοι γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο αν θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από τις, πρωτα... τις αρχικές ε, απόψεις που έχετε καταλήξει διότι αυτό θα βοηθήσει τους συναδέλφους να αποφασίσουν αν αξίζει να περιμένουν ή να κινηθούν πιο γρήγορα χωρίς να προδικάζω την απόφασή τους. Πριν από τη συνεδρίαση των συντονιστών έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον ε, εισηγητή για να μας πει αν έχει το αίσθημα ότι μετά από την υποψηνή συζήτηση προχώρησε κάπως το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε και κάτι για το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα. Σημειώνω ότι θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων στις 10 Ιανουαρίου, μια άλλη ευκαιρία για ανταλλαγή ε, απόψεων στις 10 Ιανουαρίου μετά τις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γίνει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουν συγκλίνει απόψεις μέχρι τότε και έχω και τον κατάλογο ε, ψήφων και με τις απόψεις των διαφόρων ε, ομιλητών. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε τώρα την απάντησή σας για αυτά που ακούστηκαν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω από τις γενικότητες να εστιάσω στις λεπτομέρειες. Λέγοντας εξ αρχής ότι η κατάσταση, η θέση μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Το 2008 όμως είχαμε μείον 5% ανάπτυξη όταν στην Αμερική και στην, ε, Κίνα ειδικά ήταν σύν 8%. Εμείς πηγαίναμε αντίστροφα λοιπόν. Εάν θέλουμε τώρα να έχουμε μία ευκαιρία στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να μην χάσουμε το επίπεδο ευημερίας μας και το επίπεδο της ζωής μας. Τώρα, ε, δεν συζητάμε μία τρελή ιδέα, μία παράλογη ιδέα. Ακόμα και ο καθηγητής Μόντι στην έκθεσή του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να πράξουμε κάτι για να βελτιώσουμε τη θέση μας. Δεν λέω ότι πολλές πτυχές του ζητήματος αυτού είναι περίπλοκες, αλλά όχι τόσο περίπλοκες που να μην γίνονται κατανοητές από τους εμπορευόμενους και τους καταναλωτές. Γι' αυτό θα αναφερθώ σε ορισμένες ε, λεπτομερείς παρατηρήσεις που έγιναν. Σωστό είναι να καλυφθούν τα ψηφιακά προϊόντα σε όλα τα κεφάλαια πλην του κεφαλαίου 4. Οι ειδικοί στην προστασία καταναλωτών λένε ότι η ρύθμιση για τα ψηφιακά προϊόντα πρέπει να είναι στεγανή, να μην έχει παραθυράκια. Είναι υπηρεσία ή είναι εμπόρευμα. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Είχαμε και μία έκθεση από εμπειρογνώμονα και πάλι δεν συμφωνήσαμε. Τώρα, εάν η Κομισιόν θέλει σε τέσσερις μήνες να προτείνει πάλι κάτι άλλο, τότε θα πρέπει να προσέξουμε να μην ενσωματώσουμε, όπως είπε και ο κύριος Λέχνερ, κάτι για τα ψηφιακά προϊόντα σε αυτή την οδηγία, εάν σε τέσσερις μήνες έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν επιφυλάξεις, αλλά δεν θέλουν και κάθε δύο εβδομάδες να κάνουν μια προσθήκη στο αστικό τους δίκαιο. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα των ψηφιακών προϊόντων. Όσον αφορά τη μελέτη επιπτώσεων που είπε η κυρία Βάιλερ, συμφωνώ μαζί, σου, μαζί σας. Στις 18 Νοεμβρίου όμως είδαμε και τη μελέτη επιπτώσεων της Κομισιόν επί μιας εκθέσεως. Εάν έχουμε τώρα και άλλα παρόμοια αιτήματα για μελέτη επιπτώσεων στις τροπολογίες θα μπορέσουμε και αυτό να το συζητήσουμε. Επίσης ευχαριστώ τον κύριο Λέχνερ που είπε ότι ο τελικός μας στόχος είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουμε να είναι εφικτά και εφαρμόσιμα. Γι' αυτό ακριβώς το άρθρο 2α πρότιμα πρότεινα να καλύψουμε μόνο τέτοιες συμβάσεις που να συμπεριλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών και όχι συμβάσεις οι, οι οποίες ε, κλείνονται στη... στην πόρτα όταν χτυπά κάποιος το κουδούνι θέλουμε να, για να μας πουλήσει ας πούμε τζάμ, διπλά τζάμια. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να καλυφθούν ακριβώς οι συμβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν και να καλυφθούν νομοθετικά. Πιστεύω ότι από τα κεφάλαια 1-2 μπορούν να εφεληθούν και οι καταναλωτές και η εσωτερική αγορά. Το ερώτημα είναι το κεφάλαιο 4 τι θα μας προσφέρει Είμαι πρόθυμος να συζητήσω με τους συναδέλφους και να καταλήξω σε σωστούς συμβιβασμούς. Ό,τι είπε ο συνάδελφος τώρα Χουανόκ. Και εκεί δεν διαφωνώ, συμφωνούμε. Στο άρθρο 5 θέλουμε να εδραιώσουμε γρήγορες ε, διαδικασίες επικοινωνίας, τηλεπικοινωνιών δηλαδή, και όταν έχουμε μέγιστη προθεσμία 30 μέρες οι συμβαλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν τι θέλουν. Αν δεν συμφωνήσουν τι θέλουν τότε θα ισχύουν οι 30 μέρες. Σε πολλά αστικά δίκαια κρατών μελών ήδη έχει ενσωματωθεί αυτή η διάταξη. Επανέρχομαι στην κυρία Γκέπαρτ. Ε, κατανοώ όσον αφορά τις παρατηρήσεις σας για τα μέσα, τους τρόπους πληρωμής. Υπάρχει μία πρόταση τη 1132 και 1135 που αναφέρονται συστήματα πληρωμών. Από τις δύο αυτές τροπολογίες προσπάθησα εγώ να συντάξω μία συμβιβαστική. Οι δύο αυτές προέρχονται από τη σοσιαλιστική ομάδα. Έχουν καλή πρόθεση, δεν λέω, αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Είμαι, έχω μία ανοιχτή προσέγγιση, αλλά στο τέλος Εάν κολλήσουμε σε κάθε λεπτομέρεια, θα χάσουμε το δάσος από τα πολλά δέντρα. Γι' αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο Ροσφόρ που λέει ότι σε κάθε διαδικασία τέτοια που ξεκινάμε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν η βασική οδηγία έχει διευρυνθεί, έχει απλωθεί υπερβολικά και μήπως θα πρέπει να επανέλθουμε στο βασικό σκελετό πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν μαζί με πολλές επικοδομητικές τροπολογίες μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις. Όμως, εάν κολλήσουμε σε τροπολογίες τόσο ειδικέ όσο αυτές των δύο συναδέλφων και αρχίσουμε και μπλέκουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε συμβιβασμό. Γι' αυτό λέω, Ευχαριστώ όλους για την υποβολή τροπολογιών. Με το υλικό που έχω στα χέρια μου θα προσπαθήσω να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουμε και πιστεύω ότι στις συζητήσεις που θα κάνουμε με τους κοιόδης εισηγητές και στις συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας θα προχωρήσουμε. Απλά δεν είναι τα πράγματα, αλλά δεν είναι και αδύνατα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνω μια έκκληση στην καλή διάθεση όλων των συναδέλφων και σε όσους έκαναν εξαιρετική εργασία προετοιμάζοντας ε, την, ε, τις τροπολογίες και ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε μια, ε, ένα εύρος συζητήσεων με την αναβολή της ψηφοφορίας και θα δούμε πού βρισκόμαστε στις 26 Ιανουαρίου για τελευταία φορά πριν ψηφίσουμε στις 27. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να συνεισφέρει κάτι ακόμα στη συζήτηση. Ναι. Ήθελα να κάνω μία παρατήρηση ε, ακόμα, διότι είναι ένα από τα σημεία στα οποία διαφωνούμε. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε πλήρη εναρμόνιση στο κεφάλαιο 4 ή όχι. Εάν θέλετε σε ορισμένα σημεία να επιτύχετε πλήρη εναρμόνιση, θα πρέπει να δεχτείτε ότι θα υπάρξει ένας τεράστιος κατάλογος, ευρύτατος. Εάν δεν θέλετε να επιτύχετε πλήρη εναρμόνιση, τότε, παραδείγματο χάρη, στα συστήματα πληρωμών, στα μέσα πληρωμών, μπορούμε να επιτύχουμε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Ο συμβιβασμό τον οποίο προτείνεται είναι καλός. Εκτός από την τελευταία πρόταση που λέτε ότι πρόκειται για πλήρη εναρμόνιση. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε περί ποιων μέσων ε, συστημάτων πληρωμών ε, ομιλούμε. Ποια είναι αυτά τα συστήματα. Ε, μπορεί κάποιος να σκεφτεί άλλη έναν τρόπο πληρωμής. Άρα λοιπόν πώς θα καλύψουμε, πώς θα μπορέσουμε ποτέ να καλύψουμε πλήρως και να εναρμονίσουμε πλήρως όλους τους τρόπους πληρωμής σε όλε τις χώρες με όλα τα προϊόντα. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ρεαλιστικό. Υπάρχουν ε, και τα απολωλώτα πρόβατα, τα, τα, οι οποίοι προσπαθούν να παρανομήσουν. Υπάρχουν πάντοτε οι επιτίδοι, οι οποίοι θα βρουν έναν άλλο τρόπο πληρωμής που δεν τον έχουμε σκεφτεί εγώ και θα παρακάψουν τη δική, τη δική μας προστασία. Λοιπόν, μην ξεχνάμε και αυτούς, τους απαταιώνες. Θέλετε να έχετε τελευταία λέξη κύριε Σουάμπ. Ναι. Εντάξει. Πολύ σωστή η παρατηρήσή της κυρίας Γκέπαρτ. Γι' αυτό πιστεύω ότι το κεφάλαιο 4 θα πρέπει να παραμείνει στη βάση της ελάχιστης εναρμόνισης. Αναφέρθηκα στο άρθρο 22 για τις παραδόσεις και το είδος του ρίσκου που αναλαμβάνουμε. Υπάρχουν 26 κράτη-μέλη τα οποία έχουν διευθετήσει το θέμα του ρίσκου. Σε ένα κράτος μέλος η κατάσταση είναι σαφής. Το αργότερο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούμε να, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία είναι στιγμή όπου το προϊόν είναι στα χέρια του παραγγέλλοντος. Υπάρχει λοιπόν μόνο ένα κράτος μέλος όπου αρχίζει η διαδικασία της ανάληψης ε, ρίσκου πριν γίνει η παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή. Ε, πρέπει να καταλήξουμε ποιο θα είναι το κατάλληλο χρονικό στη, στη σημείο όπου θα ξεκινήσει η ανάληψη ευθύνης. Ε, πριν από την παράδοση ή μετά από την παράδοση. Είμαι, έχω ανοιχτή προσέγγιση, η δική, μου, ε, η δική μου πρόταση είναι να εφαρμόσουμε ελάχιστο επίπεδο εναρμόνηση στο κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 4. Να είμαι ξεκάθαρο. Ελάχιστη εναρμόνιση, δική μου πρόταση. Εάν συμφωνείτε με αυτό, τουλάχιστον θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Το ερώτημα ήταν, στις 9 Δεκεμβρίου, αυτό είναι η τελευταία μου παρατήρηση, στις 9 Δεκεμβρίου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις δημοσιονομικές πτυχές και στην χρηματοδότηση ορισμένων διαδικασιών και επίσης στον τομέα τη πληροφόρηση. Εδώ θα ήθελα που καταφέρουμε να συζητήσουμε και για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο. Και εφόσον επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε κάποιους τομείς εναρμόνισης που προτείνεται, θα ήταν σκόπιμο να τους υπογραμμίσουμε αυτούς τους τομείς με ένα σύντομο σημείωμα που θα απευθύνεται στους συναδέλφους. Πάντως, κάποια πρόοδο σημειώθηκε. Θα, έχουμε περαιτέρω συζήτηση σε 9 Δεκεμβρίου και θα, μια ενημέρωση για τις προόδους που έχουν σημειωθεί για να δούμε πού έχουμε φτάσει από πλευρά συμβαστική λύση. Και κατόπιν στις 10 Ιανουαρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε, ελπίζω, τα ε, τα προβλήματα που εναπομένουν για να πάει το κείμενο για ψηφοφορία στις 26 Ιανουαρίου. Φοβάμαι ότι θα χρειαστεί πολύ να δουλέψει στη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Επιτροπή. Uh, να πιω μια γουλιά γιατί πνίγηκα και συνεχίζω. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της ε, δημόσιας συνεδρίασής μας. Αύριο το πρωί, σας θυμίζω, θα ξανασυναντηθούμε στι 9. Θα γίνει μια ψηφοφορία στις 10. Εκθέσεις, ε, για τις δύο εκθέσεις και μετά θα συνεδριάσουμε μέχρι το μεσημέρι και κατόπιν αύριο το απόγευμα. Οι συντονιστές, εάν είστε σύμφωνοι, να αρχίσουν, να αρχίσει η συνεδρίασή τους στις 5 και 20 για να έχουμε